ίσης ψήφου. Σε μισό λεπτό βεβαίως. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφους για την έκθεση Για ένα λεπτό. Η κυρία Κιούνε. Ένα λεπτό. Κυρία Κιούνε. Έχετε το λόγο, κυρία Κλούνε, για ένα λεπτό, για να εξηγήσετε την ψήφο σας. Ε, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω το στόχο του να έχουμε μία και μόνη υπηρεσία στην Ευρώπη για να απλουστεύσουμε τα ταξίδια στην Ευρώπη, στην ενιαία αγορά. Οι επιβάτες θα μπορούν να αγοράζουν και να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους στο μέλλον. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε τα ταξίδια ε, με συνδυασμένες μεταφορές. Πρόκειται για μια πολύ περιπλοκή διαδικασία το να αγοράσουμε αεροπορικά, ε, εισιτήρια, συνδρομικά εισιτήρια κτλ. Με ένα και μόνο εισιτήριο θα πλουστεύσουμε το σύστημα και το σύστημα θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Και επιπλέον ε, το σύστημα μεταφορών θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, φιλικό προς το χρήστη. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα ε, Ταξιδιών θα είναι πολύ καλύτερη και κανένας θα μπορεί να σχεδιάζει πολλαπλά ταξίδια, ε, θα έχει καλύτερες ευκαιρίες ως καταναλωτής αλλά και ως τουρίστας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όσοι αποχωρούν από την αίθουσα λίγο πιο ήσυχα. Η κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ίδρυση και η εφαρμογή ενός συστήματος ε, πολυτροπικών ε, εισιτηρίων με μία ενιαία έκδοση στην Ευρώπη θα διευκολύνει όχι μόνο τους επιβάτες, αλλά θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα και να προωθήσουμε την ανάπτυξη για όλο τον τομέα. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με κάπως ασαφείς στόχους που τύφονται σε ό,τι αφορά την σύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε ό,τι αφορά το 2020 και σε ό,τι αφορά τους διάφορους τρόπους ε, μετακίνησης και ταξιδίου. Δεν μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν με το στόχο του να τεθούν τέτοια πρότυπα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες και την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων και πιστεύω ότι αυτό θα σήμαινε απώλεια ε, επιχειρηματικών ε, ευκαιριών για πολλές εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σεϊμούρ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, και πάλι βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα αυτή να μιλάω κατά διαφόρων σχεδίων έκθεσης ε, και ψηφίσματων. Καλή αυτό το ψήφισμα να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα έκδοσης συντηριών. Ο λαός στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να υπάρχει μια βάση δεδομένων από το υπερκράτος το ευρωπαϊκό που θα αποθηκεύονται τα στοιχεία τους. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν είναι χαλασμένο. Το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων μας είναι μια χαρά όπως έχει. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε μόνοι μας, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι η κυβέρνηση της ε, του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει τεράστιε περικοπέ και δεν μπορούμε να σπαταλάμε χρήματα σε τέτοιου τομεί. Είναι ανέφικτο να πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί και πρέπει να αλλάξει ο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα κάτοικο στο χωριό ε, τη ε, αγγλία ε, τον τρόπο που εκδίδεται δικά του. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί να αλλάξουμε το σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Άντερσον την οποία δεν τη βλέπω. Περνάμε στον κύριο Μαμίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, γιατί το ολοκληρωμένο σύστημα εισιτηρίων είναι πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ολοκληρωμένο και καλά διαρθρωμένο σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τις χώρες που δεν είναι καλά συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες χώρες. Η χρήση των μοντέρνων και σύγχρονων τεχνολογιών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών και θα προωθήσει την ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία και το Κοινοβούλιο την υποστήριξε. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Κύριε Κόρβιν, ε, ζητήσατε να... το λόγο για να κάνετε επεξήγηση ψήφου. Αν ναι, έχετε το λόγο τώρα. the time about the Μιλάμε για την ποικιλομορφία. Το κοινοβούλιο μας υποτίθεται ότι υποστηρίζεται την ποικιλομορφία αλλά στην πραγματικότητα ψηφίζουμε για την ε, ομοιομορφία των πάντων. Δεν ψηφίζουμε την πολυμορφία, αλλά την ομοιομορφία. Τώρα το κάνουμε αυτό μέσω των, ε, του ενιαίου αυτού εισιτηρίου. Η κυρία Άντερσον έφτασε, της τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι Λονδρέζα και Βρετανίδα βουλευτής. Έχω άθλιες σκέψεις σε σχέση με την ε, τραγωδία που συνέβη δέκα χρόνια πριν και ανάγκασε όλες τις κοινότητες στο Λονδίνο να συνεργαστούν και τους ε, εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών. Σε σχέση με τα εισιτήρια, θα ήθελα να σας πω ότι καλωσορίζω την έκθεση για τα εισιτήρια και υπερψήφισα τις ε, συστάσεις. Θέλω να υπογραμμίσω την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στους σταθμούς τρένου, στα σημεία αλλαγής, στους κόμβους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι να μπορούν να ταξιδεύουν. Επίσης, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά προς το συμφέρον και το καλό όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έκθεση Νίκολσον για την εφαρμογή του πακέτου γάλακτος. Ε, ο λόγος στην κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό. Κυρία Χάρκιν. Υποστήριξα αυτή την έκθεση του Jim Nicholson. Έρχεται μια κέρια στιγμή. Έχουμε 634, ε, λιγότερο τα μισά από ό,τι είχαμε το 2014. 16% κάτω από το χαμηλότερο σημείο του που ήταν το 2009. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά. Ε, αυτό ε, σημαίνει ότι 35.000 ευρώ το χρόνο χάνει ένα, ο μέσος ε, κτηνοτρόφος Ιρλανδός. Όλα πηγαίνουν ε, προς τη λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω θερμή υποστήριξη στο Κοινοβούλιο για να πούμε ότι το σημερινό ε, δίκτυο ασφαλείας, η ιδιωτική αποθεματοποίηση και η δημόσια στήριξη δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε ε, την αστάθεια που υπάρχει και οποιαδήποτε κρίση στον ε, γαλακτοκομικό τομέα. Θα ήθελαμε να, η Κομισιόν να, είναι πιο, να τίνει πιο ευηκοούς και η τιμή παρέμβασης θα πρέπει να ε, αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές τιμές αγοράς και την απώλεια σε αυτές και στην παραγωγή. Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο κοστίζει η παραγωγή του γάλακτος και πόσο ε, κερδίζουν οι κτηνοτρόφοι. Ε, στην πραγματικότητα θα πρέπει οι αγορές να εξυπηρετήσουν τους, τον κόσμο. Ας πούμε την αλήθεια ως ευρωβουλευτές. Και με αυτέ τις πολιτικές νομίζω ότι σκοτώνουμε τον κάμπο και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πλήρη ε, επισητιστική ασφάλεια. Πρέπει να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι τόπου για να μπορέσουν να επιβιώσουν κάθε μέρα. Γιατί το να σκοτώνουμε τον κάμπο, τον κάμπο σημαίνει ότι σκοτώνουμε τον εαυτό μα, Αυτό είμαστε. Ε, μας κλέβουν την ταυτότητά μας σε αυτό το κοινοβούλιο. Ίσως δεν είμαστε η πλειοψηφία, αλλά το ρυθμό, τον παλμό της ιστορίας τον καθορίζουν οι άνθρωποι. Ε, και στην πραγματικότητα εδώ οι μεγάλοι ε, κερδοσκόποι κερδίζουν και χάνουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι τι κάνουν οι λαοί. Όταν δεν έχουμε μνήμη, χάνουμε. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ με το πέρασε των ποσοστώσεων μετά από 30 χρόνια για το γάλα έχουμε μια πελώρια πρόκληση για την βιομηχανία αλλά και μια ευκαιρία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και υπήρξαν θετικές αντιδράσεις στην Ιρλανδία όπου η κτηνοτρόφοι προσπαθούν να αναβαθμίσουν και να επενδύσουν σε αισθήματά τους για να αυξήσουν, ε, να εντετικοποιήσουν την παραγωγή. Με χαρά υποστήριξα την έκθεση διότι μεταξύ άλλων αναγνωρίζει τη σημασία του γαλακτοκομικού τομέα για τις εξαγωγές ε, και για εγχώρια κατανάλωση, αλλά κυρίως για τις εξαγωγές ε, και επίσης πραγματεύεται και τα μέτρα για την εφαρμογή για να αντιμετωπιστεί και η πτυτικότητα των τιμών ε, που ε, συνιστά μεγάλη ανησυχία για τους ε, γαλακτοπαραγωγούς κτηνοτρόφους. Νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρη η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι υπάρχει έλλειψη σιγουριάς και ασφάλειας για τους κτηνοτρόφους και εκείνοι προσπαθούν από την πλευρά τους να επενδύσουν. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια θετική παρέμβαση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. κύριος Μπόγκοβιτς. Με το πέρας των ποσοστώσεων μειώθηκαν κατακόρυφα οι τιμές και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ο κλάδος. Αυτό προφαίνεται και από την έκθεση Νίκολσον. Εγώ Είμαι από τη Σλοβενία και η γαλακτοπαραγωγή είναι ο βασικός μας τρινοτοφικός τομέας. 60% περίπου της γης είναι βοσκοτόπια και Έχουμε πολλές ε, ορεινές περιοχές όπου ε, δυσχεραίνεται η παραγωγή, είναι δύσκολες οι συνθήκες ε, και όταν είναι τόσο χαμηλές οι τιμές νιώθουν πολύ μεγάλη πίεση οι κτηνοτρόφοι, κυρίως όταν είναι ευμετάβλητες οι τιμές όπως τα τελευταία χρόνια. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει την κατάσταση, να δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, ούτως ώστε οι γαλακτοπαραγωγοί να μπορέσουν να επιζήσουν για να αυξηθούν και οι εξαγωγές και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των προϊόντων. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νέκοφ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα μέτρα που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επαρκούν. Δεν αντιστοιχούν στην πρόκληση ε, στην οποία καλύτερα να επεξέλθουν οι παραγωγοί γάλακτος, ε, γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Ρωσία πριν από λίγες ημέρες ανανέωσε το εμπάργκο ε, για τις εισαγωγές γάλακτος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη απογοήτευση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μηχανισμοί που προτάθηκαν ε, πέρυσι απεδείχθησαν ανεπαρκείς ε, ενώπιον του εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε επίσης τα διάφορα μέτρα που σχετίζονται με τα διάφορα είδη τυριών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλείται να διευρύνει να, τον κατάλογο των προϊόντων, κυρίως για τα τυριά, και να αναθεωρήσει διάφορα μέτρα σε αυτό τον κλάδο. Λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Χρειάζεται παρέμβαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε, κύριο Μαμίκιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε και ψήφισα για την έκθεση αυτή, γιατί στις 31 Μαΐου του 2015 οι του γάλακτος καταργήθηκαν και η Ρωσική Ομοσπονδία επέμβαλε μπάργκο στα γαλακτοκομικά προϊόντα και αυτό έπληξε ιδιαίτερα τους Λετωνούς ε, ε, γεωργούς και έπεσαν τα έσοδα για τι πραγματικές οικογένειες, όχι για δείκτε. Δεν μιλάμε για δείκτε και αριθμητικά στοιχεία, μιλάμε για πραγματικές οικογένειες που διακυβεύεται η επιβίωσή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βοηθηθούν οι βαλτικέ χώρες και οι άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του παραγωγού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι... Nous allons donc passer aux explications de vote sur le rapport de Monsieur Πάμε στην έκθεση Σαραντήλη. Ο εξωτερικό αντίκτυπο εμπορική και επενδυτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτε χώρε. Ε, ο κύριο ε, Μάμικιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή γιατί η συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για να πετυχθούν οι στόχοι της ε, μείωσης της στόχας. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των χωρών αυτών και να μην δρούμε βάσει ενός ξεχωριστού οράματος. Σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλουμε project γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα για τους κατοίκους της ε, εκάστοτε χώρα και σε τελική ανάλυση αυτοί δεν ενδιαφέρονται γιατί μόνο οι πόροι τους ενδιαφέρουν και έτσι τα έργα αυτά παραμένουν ανεφάρμοστα. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε όταν μιλάμε για τέτοια έργα σύμπραξη δημοσίου. Σας ευχαριστούμε. Έτσι, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Τη δεύτερη ημέρα της Ολομέλειας αγωνίστηκα για να το πετύχω. Ευχαριστούμε. Ο πόλεμος κατά αυτών των συμβουλών ναι, και των προβλημάτων που δημιουργούν είναι ένα από τα βασικά προβλήματα στην Αγγλία. Δηλαδή, ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολλά ε, νοσοκομεία στη, στην περιφέρειά μου και σε άλλες ε, φτωχοποιημένες περιοχές ε, της Αγγλίας έχουν αυξηθεί τα τέλη για αυτούς που θέλουν να πάνε να παρκάρουν στο νοσοκομείο για να πάνε ε, να, να δούνε τους συγγενείς τους. Θέλουν να περάσουν απλώς για να περάσουν να πάνε ε, να περάσουν από τους δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν στο νοσοκομείο και να επισκεφτούν τους εγγενείς τους. Πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτά τα οδικά τέλη. Ευχαριστούμε και τώρα ε, ψήφων για την έκθεση μέλο κ. Μπόκοβιτς για τον τομέα των απορρικυπευτικών και τη μεταρρύθμιση του 2007. Ε, ευχαριστώ. Υποστήριξα την έκθεση μέλο διότι οι οργανώσει παραγωγών στον τομέα των απορροκυπευτικών είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην περικοπή του κόστους και στο μάρκετινγκ σε αυτές τις δυσχερές συνθήκες στον τομέα της γεωργίας. Μόνο το 1 τρίτο της αρρώσιμης γης αντιστοιχεί στα απορροκυπευτικά και η παραγωγή ε, ανέρχεται στο 18%. Είναι εντατική δηλαδή η παραγωγή και έχουμε 550.000 θέσεις εργασίας. Εξεκάθαρα μέσα στην έκθεση βλέπουμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχουν οργανώσεις παραγωγών. Στη χώρα μου στη Σλοβενία δεν υπάρχουν τέτοιες Έβαλα τα δυνατά μου για να διοργανώσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια διάσκεψη, τόσο ώστε να εμπνευστούμε από τις βέλτιστες πρακτικές του Βελγίου, παραδείγματος χάρη. Ελπίζουμε ότι ο Σλοβαίνος υπουργό με τις νέες εξελίξεις θα καταρτήσει στρατηγική και θα συστήσει τις πρώτες οργανώσεις που παραγούν. Ευχαριστούμε κύριο Νίκο. Υποστηρίζω ολόθερμα την παράφο 18 της έκθεσης για τα προκυπευτικά και κυρίως την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδώσει οικονομική βοήθεια ε, για τις νέες οργανώσεις παραγωγών προκυπευτικών. Αυτές οι οργανώσεις είναι ισχυροί μηχανισμοί στα χέρια των παραγωγών τη στιγμή που διαπραγματεύονται με, τις υπο... με τους υπόλοιπους ε, συμμετέχοντες στην αλυσίδα ε, παραγωγής. Και είναι ε, πολύ δημοφιλής στις ε, καινούριες χώρες όπως η Βουλγαρία. Οι, ανα... οι εξελίξεις της περσινής χρονιάς και κυρίως το ρωσικό εμπάργο, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ανεπαρκή. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει επιπλέον πόρους άμεσης βοήθειας προς τους παραγωγούς, αντί να αφήσει τους παραγωγούς που είναι εκατομμύρια χωρίς καμία προοπτική και χωρίς ψωμί στο πιάτα τους. Θα ήθελα να ξεκίνησε και μια προπαγάνδα ε, μεταξύ των νέων ε, για να τους δείξετε ότι μπορούν να κερδίσουν μέσω της γεωργίας ε, τη ζωή τους. Βεβαίως απομονωμένες περιοχές, οι ορεινές περιοχές ε, είναι πολύ ε, ε, προβληματικές και συχνά πρέπει να κάνουμε κάτι. Σταματάει εδώ η σύνοδος και ξαναρχίζουμε στις 3 η ώρα.